από την 7η Απριλίου 2014 την έλαβε υπόψη και καλωσορίζω τη νέα ή παλαιότερη συνάδελφο και υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ευρωκοινοβουλίου του Κανονισμού κάθε μέλος συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στα, στις συνεδριάσεις ε, του Ευρωκοινοβουλίου εφόσον δεν έχει υπάρξει κάποια ένσταση και υπό την προϋπόθεση ότι η κυρία Σάξα έχει δηλώσει ότι δεν έχει κάποιο αξίωμα το οποίο να